από εκείνου που είναι πάντα εδώ και θα κοιτάξω να, καθισ... να κολλησιεργήσω λίγο μέχρι να έρθει η κάρτα. Γραπτή δήλωση 007, όχι, όχι, συγγνώμη. Γραπτή δήλωση 0007 του 2012 υπευλήθη από τον κύριο Μποντ, όχι, από τον κύριο Κάτσμαρετ, Μπαρία Κουτσέκ, Γκάλερ, Γκρέσ και Φάρντε Χολ για το θέμα εκπαιδευτική εργασία και ενεργός παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη. Αυτό έχει ε, συγκεντρώσει τις υπογραφές και βάσει του άρθρου 123 του κανονισμού θα ε, δοθεί στους παραλήπτες και θα δημοσιευτεί. Τα ονόματα των υπογραφόντων θα ε, συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Ο κύριος Κάτσμαρακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, για τη γραπτή αυτή δήλωση. Θα είναι σκόπιμο να την υποστηρίξετε μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάτσμαρεκ. Γραπτή 010 του 2012 για την μέρα, την εισαγωγή τη μέρα του, της μέρας του παραδοσιακού παγωτού.